Okay, colleagues, we can move on. Πρόεδρος, συνάδελφοι, προχωρούμε σε ένα σημαντικό θέμα της Επιτροπής μας. Πρόκειται για τον προγραμματισμό της Ένωσης για το 2018. Δείτε πώς περνάνε τα χρόνια. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Γκέρνς, ο οποίος παρίσταται και... Καθίστε παρακαλώ. Και ο κύριος Γκέρενς έχει τον λόγο για να μας κάνει την σχετική παρουσίαση. Προϋπολιμός 2018. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δουλειά για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να ονομαστεί επικίνδυνη αποστολή. Στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής των Προϋπολογισμών είχα την ευκαιρία να επενθυμίσω πως οι αρμοδιότητες μας ως επιτροπές, ως ε, ευρωβουλευτές είναι τέτοιες που θα πρέπει να χαρακτηριστούν από το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Και δεν ε, λεχθεί τίποτα γι' αυτό, ούτε για το Ταμείο Ανάπτυξης. Οπότε για να σας συμπληρώσω αυτή την εικόνα του background, σας προσθέτω ότι η πόρη για την αναπτυξιακή βοήθεια είναι κάτι το οποίο διεκδικείται από όλου. Υπάρχει μια ε, γενικευμένη σύγχυση. Γιατί έχουμε από τη μία την αναπτυξιακή βοήθεια, από την άλλη μεριά ε, την μεταναστευτική πολιτική. Θέλουμε να ε, εκριζώσουμε τη φτώχεια και για το μεταναστευτικό επίσης πρέπει να αφιερώσουμε κάποια χρήματα γιατί αυτό είναι πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη οπότε στην πρώτη περίπτωση μιλούμε για απόρους οι οποίοι ε, κατευθύνονται προς κάποιες δράσεις για την εκρίζωση της φτώχειας και στην άλλη περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση λέμε ότι θέλουμε να δούμε πώς πρόκειται αυτά τα χρήματα που ήταν πριν για την ψυχική βοήθεια θα πάνε εκεί που τώρα θέλουν κάποιοι άλλοι για το μεταναστευτικό. Ως γενική σκέψη μου πρέπει να σας πω ότι εδώ, όπως λέει και η φυσική, είναι κάτι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν φεύγουν α, τα χρήματα από έναν σκοπό και πάνε σε έναν άλλον, αδειάζει το πρώτο δοχείο. Δηλαδή, και με τον Brexit να δούμε τι θα γίνει, που θα χάσουμε κάποιους πόρους. Και δεν προβλέπεται τίποτα σε αυτόν τον προπολογισμό. Τι θα γίνει δηλαδή, άπαξ και αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, είναι δύσκολο να το καθορίσουμε από τώρα, αλλά από την άλλη μεριά έχουν διατυπωθεί κάποιες προτάσεις για να μπορέσουμε να ξεπράσουμε το πρόβλημα. Έχουμε πει τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις. Τελικά υπάρχει αδιαφορία. Είδατε τι έγινε όσον αφορά την συνένεση για την ανάπτυξη. Τίποτα δεν γίνεται δηλαδή δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Τίποτα δεν κάνει το Συμβουλίο. Πώς δηλαδή αυτή η δημόσια πόρη για την ε, ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο θέλουν να το σφετεριστούν τα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά. Θέλουν να κάνουν πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική, το, τη μεταναστευτική πολιτική. Πρόκειται για μια υποκρισία. Θα πρέπει αυτό να το καταγγείλουμε όταν τοποθετηθούμε για τον προϋπολογισμό. Είμαστε μόνοι μας, αλλά θα πρέπει να ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα. Τι έχουμε. Έχουμε 232 εκατομμύρια και είπαμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά τα 232 εκατομμύρια. Αν ήδη έχουν διατεθεί κάποιοι πόροι για την Τουρκία, θα πρέπει και αυτό ξεκάθαρα να διατυπωθεί. Δηλαδή πρόκειται για κάποια χρήματα που αποσκοπούν στο να λύσουν τα δικά μας προβλήματα, αλλά πάνε αλλού. Και δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη για κάποια κοινή δράση όσον αφορά τη μετανάστευση το ίδιο και για το μέσο ευελιξίας. Τι θα κάνουμε. Λίγο-λίγο θα φύγουν οι πόροι από εκεί, από την ανάπτυξη δηλαδή για να πάνε ε, στην Τουρκία επί τη βάση του σχετικού συμφώνου. Και έχουμε άλλα 20 εκατομμύρια που αφορούν ε, την ε, ανάπτυξη και αφορούν κάποιες καταστάσεις για τις οποίες δεν φταίει η Ευρώπη, δεν φταίει κάποιο κράτος μέλος, αλλά το θέμα είναι ο Τραμπ, ο οποίος ε, με τις ενεργειές του τώρα αποστερεί από κάποιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τους πόρους που χρειάζονται για να βοηθήσουν κάποιο είδου ε, ανθρωπιστική βοήθεια για τις γυναίκες σε κάποιες πολεμι, περιοχές που υπάρχει πόλεμος. Οπότε έχουμε αυτά τα 232 εκατομμύρια για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ασκήσουμε την πολιτική μας. Τι θα κάνουμε. Επίσης, το κονδύλι για την Ασία. Κατά 1,7 θα περικοπεί, αλλά και το κονδύλι για την Λατινική Αμερική. Λόγω της εφαρμογής της αρχής της διαφοροποίησης που οδηγεί τους δωρητές να περιστύλουν την ε, ενίσχυση. Ενώ θα έπρεπε να δούμε πώς θα πρέπει οι ίδιες αυτές οι χώρες να ε, βρίσκουν όλα ένα και περισσότερα χρήματα για τα προβλήματά τους. Οπότε έχουμε επίσης τη βοήθεια προς τις χώρες με διάμεσο εισόδημα και να δούμε πώς η Επιτροπή αντιλαμβάνεται την εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης σε σχέση με τον προπολογισμό. Έχουμε 14 εκατομμύρια που έχει στη θέση της η Ένωση για το 18. Και άπαξ και έχουν ε, ανακοινώσει αυτό την περικοπή των 7%. Αν αυτό γίνει, δεν έχω τώρα εδώ τα σχετικά στοιχεία. που θα οδηγήσει δηλαδή η εφαρμογή της διαφοροποίησης αλλά έχουμε εδώ αυτό το αποθεματικό και τι να σας πω, περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και να καταλήξουμε σε κάτι ε, ως γενική θέση για αυτά τα θέματα και να τα πούμε και στους άλλους τους αρμόδιους για τον προϋπολογισμό. Βασικά αυτά είχα να σας πω και όσον αφορά αυτές τις ε, γενικές σκέψεις υπάρχουν ε, τα θέματα τα οποία επανέρχονται Εντάξει, ο προπολογισμό ε, έχει ένα στενό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει αυτά να τα θέσουμε. Αυτά τα ζητήματα είναι προφανές ότι υπάρχουν ανάγκες. Και στο G7 στη Σικελία ο Ιταλός Πρωθυπουργός μίλησε για σημαντικές ανθρωπιστικές ανάγκες. Μίλησε για 7 δις ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στις χώρες που απειλούνται από την πείνα. Και έβγαλε τα ακουστικά του τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος και δεν, χωρίς να καταλαβαίνει Ιταλικά. Τα έβγαλε γιατί δεν του καίγεται καρφάκι για αυτό το πρόβλημα. Οπότε δηλαδή στον κόσμο μας σήμερα άλλοι αναλαμβάνουν τι ευθύνες τους, άλλοι υπόσχολοι θα τι αναλάβουν. Όχι, όχι η Ευρώπη. Θα πρέπει όμως η Ευρώπη τελικά να πει τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Πάλι ο δυνατός κρίκος εδώ είναι το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια γενική διαπίστωση ότι αυτό είναι πονίδιστο το πόσο τα κράτη-μέλη θέλουν να αδειάσουν τον κορβονά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτήσουν κάποιες μη ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι σκάνδαλο αυτό και θα πρέπει να το καταγγείλουμε στα πλαίσια ζήτηση για τον προπολογισμό. Σάλ, σε ευχαριστούμε και όσον αφορά το τελευταίο που είπες για την ανθρωπιστική βοήθεια. γιατί τι στην ε, Ουγγάντα και εκεί έχουμε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από το Σουδάν. Απίθυνε έκλεισε σε όλους ε, ο ΙΕ. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκριθεί και καλύψαμε 70% των αναγκών. Αλλά δεν έβαλαν το χέρι τσέπη άλλες χώρες εκτός Ένωσης. Αυτό είναι προς προβληματισμόν. Ο κύριος Νόιζα. Μετά είναι η Μαρία και μετά είναι η Αναλίζα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλώ εκ μέρους του και Παγιό, σχεδόν συγητού που δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρόν στη συνάντηση. Θα είμαι σύντομο γιατί ήδη τον Απρίλιο συζητήσαμε τον προπολογισμό να υπενθυμίσω τις πολιτικές ε, προτεραιότητες της πολιτικής μας ομάδας καταρχήν και στη συνέχεια θα μιλήσω και για τα πώς αυτά ερμηνεύονται στον προϋπολογισμό. Καταρχήν οι πολιτικές προτεραιότητες. Νομίζω ότι ο Σάγλ πάντοτε, όπως και σήμερα, είναι ξεκάθαρος για τον κανόνα του 0,7 και για την ανάγκη ε, του να αντικατοπτρίζεται στην κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα καλύψουμε το κενό το οποίο προκαλείται από την απόσυση βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια ε, κοινή ε, στάση σε αυτά τα θέματα. Τονίζουμε την πολιτική για την ανάπτυξη και την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Για την πολιτική ανάπτυξη πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εξάλληψη της φτώχειας. Θα πρέπει να, να μιλήσουμε για την ε, ανάπτυξη και για τη γεωργία και να το δούμε ως μακροπρόθεσμη επένδυση και όχι μόνο να αντιμετωπίζουμε τις άμεσες συνέπειες της φτώχειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βασιστούμε ε, στην επιτυχία μας τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα για το ICSP. Ε, Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, θα πρέπει η βοήθεια αυτή να είναι ουδέτερη και αναλογική ως προς τις ανάγκες. Μας ενδιαφέρει και πόσα χρήματα δαπανούμε, αλλά και πώς τα δαπανούμε. Και θα πρέπει να καταβάλουμε ίσες προσπάθειες ε, για να βοηθήσουμε όλους, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατά πόσο αυτό έχει σχέση με την ανταπόκριση των μέσων ενημέρωσης. Τώρα, για τον προϋπολογισμό. Περιμένουμε ακόμη τη θέση του Συμβουλίου. Μπορούμε παρόλα αυτά να κάνουμε κάποια σχόλια για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής σε κάποια σημεία είναι ικανοποιητικό όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Υπάρχουν θετικά σημεία, αλλά έχει γίνει περικοπή 7,6% στο DCI σε σχέση με το 2016. Ο προπολογισμό του περασμένου έτους καταλαβαίνουμε ότι ήταν, είχε εξαιρετικά χαρακτηριστικά γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό και να το κονδύλι για την Τουρκία. Αλλά υπάρχουν ε, συγκεκριμένα δύο γραμμές, τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουμε. Πρώτον, την περικοπή στο Εράσμους και την ε, χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να παρεμποδίζει την ε, διεθνή μας συνεργασία και την μακροπρόθεσμη επένδυσή μας στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ε, η ενίσχυση για την Αφρική δεν θα πρέπει να περικοπεί και αυτό να αποτελέσει μια ε, τάση που θα ισχύσει στο μέλλον ε, και να μην διατίθεται λιγότερα χρήματα στις χώρες της Αφρικής. Για τα πιλωτικά προγράμματα, συμφωνώ με την στάση του συντονιστού και να ακολουθήσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει. Οι προτεραιότητες με βαθμό Γ ή Δ ξέρουμε ότι σχεδόν δεν έχουν ευκαιρία να περάσουν στον προπολογισμό. Νομίζω ότι μόνο προτεραιότητες Α και Β μπορούμε να προτείνουμε. Γουατεμάλα, ε, βοήθεια για θύματα σεξουαλικής βίας, βοήθεια ε, σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείριση κρίσεων. Τέλος, Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι προς το Συμβούλιο. Τα νέα προγράμματα και προτεραιότητες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και νέα χρηματοδότηση. Χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, απλώς θα αφήσουμε νέες κρίσεις να προκύψουν όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τις τρέχουσες κρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Νόμπερτ. Δίνω το λόγο στη Μαρία Χόιμποργκ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Χάιντι Χάουτελα να παρακολουθήσει ε, τα θέματα του προπολογισμού. Δεν θα μιλήσω εκ μέρου τη, θα κάνει οι ίδια τι τροπολογίε ε, που θέλει να κάνει, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Σάρλ είπε προηγουμένω πόσο σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε τι θέσει μα στον τομέα τη ανάπτυξη και να υπερασπίσουμε ε, την πολιτική μας παλεύοντας για αυτή τον Ιούλιο του 2018, σε ένα χρόνο, θα λάβουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε δηλώσει σαφώς ποιοι είναι οι στόχοι μας για την αναπτυξιακή πολιτική. Όπως είπαμε, καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτά τα οποία ανέφερε τώρα ο Νόβερτ για την ανάπτυξη κλπ. Αν δεν ε, έχουμε παλέψει για αυτούς τους στόχους, στο επόμενο δημοπολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα καταρακωθούν αυτοί οι στόχοι. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τους στόχους μας και εγκαίρως πριν από την επόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ποια σημεία θεωρούμε εμείς σημαντικά. Βλέπουμε ότι ε, κάποια χρήματα πηγαίνουν προς τον τομέα της μετανάστευσης, ε, ξεφεύγοντας από το στόχο της ανάπτυξης και πρέπει να τα λάβουμε, τονίζω, υπόψη για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να θέσουμε τις προτεραιότητές μας να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό το οποίο θέλουμε. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια και την ειρήνη, θέλουμε σε εθνικό επίπεδο το 2% του ΑΕΠ να είναι για στρατιωτικές ε, ικανότητες, αυτό το 2% γιατί να μην το αφιερώσουμε σε ε, ανάπτυξη δυναμικού ειρήνης και ασφάλειας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μιλάμε για στρατηγικές δαπάνες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει νόημα. και η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει εγκαίρως να συζητήσει αυτά τα θέματα πριν θέσει τις βασικές γραμμές η Επιτροπή και μετά προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες μικροτροπολογίες. Εξ αρχής θα πρέπει να δηλώσουμε τους στόχους μας και η στάση της Επιτροπής να βασιστεί πάνω στους στόχους που έχουμε τονίσει ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Εγκαίρως λοιπόν να καθοδηγήσουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό και ο προπολογισμό το 2018 είναι καλή βάση για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω στο μήκο κύματο που μας είπε, που μας μίλησε τέλος πάντων ο κ. Νόιζε. Πάει το DCI στην ε, ΑΦΕΤ και άλλα προγράμματα. Επομένω τώρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, η χρηματοδότηση για το DCI θα βρεθεί εκτός προϋπολογισμού. Οπότε τέτοια θα πρέπει να είναι η γραμμή μας. Ε, προσοχή. Τι θα γίνει στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα υπάρχει DCI σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως θα πρέπει κάτι τέτοιο να μπει στην έκθεσή μας. Δεν είναι το 2% για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα. Αλλά χθε ήμουν στην Επιτροπή Προπόσμων και συζητούσαμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και θα πάνε πριν το 2020 τουλάχιστον 500 εκατομμύρια για το σχετικό κονδύλι, για την έρευνα δηλαδή την ε, αμυντική. Άρα υπάρχουν ε, χρήματα, αλλά όχι για την ανάπτυξη. Ε, γιατί λοιπόν, γιατί για όλα τα άλλα τόσο σημαντικά ε, και εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε ε, τα κονδυλιά μας. Ε, πώς να μην χρήματα. Και υπάρχει το θέμα της μετάθεσης από τον Μπαγκλαντές προς την Ευρώπη. Δεν θέλουν εκεί να κάνουν ε, περικοπές. Να, αυτό είναι παράδειγμα. Και ε, είπαμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν στο θέμα της μετανάστευσης. Σε κάποιες χώρες όμως ε, δεν μπαίνει το χέρι στην τσέπη καθόλου. Άρα θα πρέπει και εκεί να υπάρξει πίεση. Και τελευταίο, όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους, εκεί έχουμε την ε, κατάρτιση των χωρών με τις οποίες υπάρχει συνεργασία και στα σχετικά προγράμματα θα πρέπει να καλύψουμε και τα αναπτυξιακά θέματα να συζητώνται αυτά συναντήσεις ε, κορυφής. Αυτό, η κατάρτιση όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί επίσης τα σχετικά με το διεθνές εμπόριο τα θέματα των Panama Papers. Ευχαριστούμε εμείς. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μου είπαν ότι μετά το 2020 θα αρχίσει να υπάρχει χρηματοδότηση το 2018 και τέλος Φεβρουαρίου πρόκειται να εγκρίνουμε την έκθεσή μας και η Επιτροπή θα κάνει τις προτάσεις τον Ιούνιο του 2018. Επομένως και εμείς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας πριν την παρουσίαση του νέου πολιετούς πλαισίου και για τον Brexit επίσης θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην μελλοντική ε, κατάρτιση του προπολογισμού. Βλαντισλάβ και Αλμπέρτο. Ε, είναι η εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα η εκπρόσωπος της ΔΕΦΚΟ. Εμείς είπαμε ότι έχουμε τρία δις όσον αφορά τις ε, επιστώσεις ε, υποχρεώσεων και όσον αφορά πληρωμών επίσης. Είπαμε ότι όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και οι μόνες εξαιρέσεις όπως ξέρετε είναι η αύξηση της συμμετοχής του ΔΕΦΚΟ στο ISSP κατά 6,25 εκατομμύρια για το CBSD. Και επίση είπαμε θα έχουν 10 εκατομμύρια μείωση για την Αφρική που θα πάνε στο αποθεματικό και αύξηση των κονδυλίων για την ε, επικοινωνία. Το που θα δοτήσουν αυτά τα προγράμματα. Ο προπολογισμό του 2017 ήταν 2.014 εκατομμύρια, πιο πολύ από το 2018, όσον αφορά τι πιστώσει ε, υποχρεώσεων, λόγω του ότι είχαμε την τροποποιητική επιστολή, η οποία στο DCI πρόσθεσε 425 εκατομμύρια πέρσι και όσον αφορά την επικοινωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας για τη μετανάστευση και ένα από τα κονδύλια αφορούσαν την Ασία και ωφελήθηκε κατά 100 εκατομμύρια από τη σχετική αύξηση και η Λατινική Αμερική είχε περισσότερα χρήματα πέρσι γιατί υπήρχαν περισσότερα χρήματα για το καταπίστευμα της Κολομβίας, Νότιος Αφρική και εκεί συρρυκνώθηκε η χρηματοδότηση για τη συνεργασία βαθμία ε, καταργείται, η ΔΕΦΚΟ χρησιμοποίησε όσον αφορά τις υποχρέωσεις της Ένωσης για το προσφυγικό. Υπήρχε νομική, ε, ε, νομική βάση για το DCI, το, το, το Μηχανισμό Ανεψιακής συνεργασία και είπαμε ότι θα πρέπει να μην έχουμε στις πιστώσεις πληρωμών και υποχρέωσεων άλλες περικοπές με τις καινούργιες προτεραιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΚΟ. Εκπρόσωπος της ΕΚΟ. Στη, στην ΕΚΟ λάβαμε υπόψη τις αυξήσεις του προϋπολογισμού σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017. Για μας Ήδη αυτό είναι μια θετική ένδειξη ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό θα συνεχίσουμε να βοηθούμε σε Συρία και Ιράκ την κάλυψη των ε, αναγκών ε, και τι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από την πείνα, η Εμένη, η Νιγηρία, η Σομαλία και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε ε, διάφορες ε, κρίσεις εκτάκτων αναγκών και όπως βλέπετε έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα και υπάρχει αύξηση στον προϋποσμό του 2018 Σάρλ, έχεις πάλι το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου και τις επόμενες χρονιές ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν μειώσεις ε, λόγω της αρχής αυτής του χρόνου. Αλλά να μας πείτε παρακαλώ τι εκτιμάτε ότι θα ισχύσει στο μέλλον ένα αυτό. Δεύτερο. Άκουσα μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο, ο κύριος ε, Νόιζερ και ο συνάδελφος Σε σχέση και με τις δικές μου προτάσεις ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι πόροι από όσους προβλέπονται για την ανθρώπινη ανάπτυξη. αυτό σαν τοποθέτηση έναντι των θέσεων Τραμπ το έρασμος συν θα πρέπει να ξαναγυρίσει στα προηγούμενα επίπεδα και όσον αφορά την μετακίνηση των πόρων από την αναψυχική βοήθεια σε άλλες ε, πολιτικές της Ένωσης που είναι άσχετες με την ανάπτυξη. Είπαμε για άμυνα και μετανάστευση. Ε, εκεί θα πρέπει να έχουμε μία ξεκάθαρη σκληρή θέση. Κύριε Νόιμπερτ μας μίλησε για παρακολούθηση στενή ε, του θέματος, για αυτό το 2% που αφορά το, τα μέλη του ΝΑΤΟ που είναι μέλη της Ένωσης και τα σχετικά με την άμυνα. 2%. Αυτό σημαίνει για τις περισσότερες χώρες διπλασιασμό των δαπανών. Εάν τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν διπλάσια από όσα δίνουν τώρα στην ε, αναπτυσιακή βοήθεια, ή τα δώσουν τώρα στην άμυνα, και αυτό είναι μία υπόσχεση που δεν μπορεί να τηρηθεί, γιατί μιλούμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα χρηματοδοτήσουν τα υπόλοιπα, αυτό να τους ρωτήσουμε. Αφού δεν υπάρχουν τώρα χρήματα. Γιατί για να υπάρξει το Ταμείο Άμυνας χρειάζονται κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν. Άρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λένε. Θα πρέπει να έχει αποφασιστική τοποθεσία το Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να μας βοηθήσει και η Επιτροπή χωρίς καμία επιφύλαξη. Γι' αυτό θα πω στην να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε οι πιστώσεις να μην περικοπούν καθόλου. συνεργάτες μου θα είναι σε συνεχή επαφή με τη γραμματεία μας και με τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες και έτσι να έχουμε προτάσεις συγκεκριμένε που έχουν συγκεκριμένα ποσά για τον προϋποσμό του 18. Σε ευχαριστούμε, Σάρλ, πρώτος, για τις τροπολογίες στην ΔΕΒΕ. Έχουμε 18 Ιουλίου, θα ψήσουμε 30 Αυγούστου και θα συζητηθεί το σχέδιο που θα ψηφιστεί στις 25, 25 Αυγούστου. Α, συγγνώμη που ε, έχασα αυτή την σημαντική συζήτηση και συγγνώμη ε, γιατί άργησα, αλλά θέλω να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε ο Σαλ Γκέρενς, ότι θα πρέπει η Επιτροπή μας να εξασφαλίσει ότι οι πόροι για την ανάπτυξη δεν θα περικοπούν. έχει αποδυναμωθεί η νομική βάση με αυτό το ε, μέσο της άμυνας, ασφάλειας κλπ. Γιατί ακριβώ θέλουν την αναψιακή βοήθεια να την ε, αποστερήσουν από ε, του, του, τους πόρους. Και αύριο να δούμε τι θα πει η νομική υπηρεσία. Αυτά που θα κάνουν δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Και θα υπάρξει και κάποια γνωμοδότηση νομική προς την Επιτροπή. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα το ξανασυζητήσουμε τέλος Αυγούστου που θα γίνει η ψηφοφορία για τις τροπολογίες. Τελειώσαμε νωρίς αυτό το θέμα. Το επόμενο είναι ε, θέμα που θα ζητηθεί από κοινού με την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σε σχέση με την κατεπίγουσα βοήθεια προς την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα εκείνο γιατί τέλος του μηνός έχουμε περικοπή των πόρων της ΕΚΟ. Και θα υπάρξει έτσι κενό στη χρηματοδότηση, όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και υπάρχει αυτό το θέμα του πώς θα εξασφαλιστούν οι βασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Στις 11 θα ξαναρχίσουμε, οπότε και μέχρι τότε διάλειμμα. Ελπίζω να έρθουν σε της Επιτροπής ε, Τους έχω ειδοποιήσει. Ελπίζω θα έρθουν. Θα τα πούμε στις 11. Α, ναι, ναι. Κοιτάξτε, μετά έχουμε το θέμα της Ερυθρέας. Εδώ γιατί το πολύ να έχουμε τελειώσει με το επόμενο θέμα για να μπορούμε να έχουμε διερμηνείς για την Ερυθρέα μετά.